Good morning everybody. Please... Uh, Καλημέρα σας. Παρακαλώ καθίστε. Καλώς ήρθατε στη σημερινή μας συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών. Ακόμη δεν έχω αποφασίσει αν θα μιλήσω αγγλικά ή σουηδικά. Ξέρω ότι είναι εξαιρετική η διερμηνία σήμερα. Παρακαλώ λοιπόν συνηθίστε την σουηδική γλώσσα γιατί θα τη χρησιμοποιώ που και που. Μπορεί να λέω να μιλάω αγγλικά και μετά κάποια στιγμή να ε, το γυρίσω στα σουηδικά. Είναι η πρώτη ε, πλήρης ε, συνεδρίαση της οποίας προεδρεύω σήμερα. Χαίρομαι πολύ που είστε τόσοι πολλοί. Είναι εδώ εμπειρογνώμονες, η γραμματεία, η νομική υπηρεσία και θα ήθελα να κηρύξω την έναρξη της σημερινής μας συνεδρίασης και να σας ζητήσω να εγκρίνετε την ημερήσια διάταξη. Μπορώ να θεωρήσω ότι εγκρίνετε. Ωραία. Ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα τι αποφάσει των συντονιστών. Μία ολόκληρη ώρα περάσαμε με τους συντονιστέ. Καταρχάς ορίσαμε εισηγητή για την ε, ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων ε, του διαμεσολαβητή. Ε, θα την αναλάβει ο κύριος Βαλένσα. Επίσης θα έχουμε την κανονική διαδικασία διορισμού ε, ορισμού ε, σκιωδών εισηγητών. Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να υποβάλλετε στη γραμματεία τα ονόματα των σκιωδών εισηγητών εντός μιας εβδομάδας. Δεύτερο, δεύτερος ε, εισηγητής δραστηριότητες για το 2014 στην ε, ομάδα των σοσιαλιστών. Ε, δεν γνωρίζουμε ακόμη ε, το όνομα των, του εισηγητή, ούτε των σκιωδών εισηγητών. Τώρα, η δικτυακή πύλη, τι, το συζητήσαμε, είπαμε ότι την Παρασκευή θα έχουμε μία συνεδρίαση, μετά θα πατάμε το κουμπάκι και θα πηγαίνουν τα σχετικά στοιχεία εκεί. Μιλήσαμε επίσης για την ανεπιτυχή πρωτοβουλία των πολιτών, ε, για τις ανεπιτυχείς πρωτοβουλίες που δεν συμπληρώνουν τον αριθμό των 1 εκατομμυρίου υπογραφών από 7 διαφορετικά κράτη-μέλη. Είπαμε όμως ότι μπορεί να τους καλέσουμε για ε, μία ακρόαση εδώ στην Επιτροπή μας. Είπαμε ότι κατά περίπτωση θα αποφασίζουμε. Δεδομένου ότι τώρα ε, ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας, έχουμε πάρα πολύ οργάνωση ε, μπροστά μας, πρέπει να οργανωθούμε με την γραμματεία και δεν θα έπρεπε να αναλαμβάνουμε πάρα πολλές πρωτοβουλίες για την ώρα. Μετά περάσαμε στο προγραμματισμό των ακροάσεων του 2014 ε, που πρέπει να τις υποβάλουμε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Οι ομάδες πρέπει γραπτός να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη γραμματεία. Στη συνέχεια κάναμε μια συζήτηση για το έγγραφο προβληματισμού που σας έχω αποστείλει. Ήταν μια καλή και επικοδομητική συζήτηση είχα την εντύπωση ότι, ότι άρεσε στους συναδέλφους η δουλειά που έκανα το καλοκαίρι. Όσον αφορά τώρα τα εκρεμή, τις εκρεμείς επισκέψεις της διερευνητικού χαρακτήρα, αποφασίσαμε ομοφόνος στην συνάντηση των συνεδρίων των συντονιστών τον Ιούλιο να τις ξανασκεφτούμε γιατί έχουμε πάρα πολλή δουλειά ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί πολύ, μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον και επικοδομητικό το να κάνει κανείς τέτοιες επισκέψεις, αλλά πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2015 και σας καλούμε βεβαίως ε, και πάλι γραπτός να υποβάλλετε τις προτάσεις σας το συντομότερο δυνατόν. Όσον αφορά την εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή θα γίνουν δημόσιες ακροάσεις στις 2 Δεκεμβρίου. Η εκλογή θα γίνει τον Ιανουάριο του 2015 κατά την Ολομέλεια, της Συνόδου Ολομέλειας στο Στρασβούργο. Εμείς, η Επιτροπή Αναφορών, ε, θα οργανώσουμε την ε, ακρόαση, θα είναι ανοιχτή στα μέλη ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει του κανόνα 219 και όπως γνωρίζετε έχουν ε, συλλέξει, ε, έχουν συλλέξει συνάδελφοι υπογραφές ε, για να υποστηρίξουν έναν συγκεκριμένο υποψήφιο. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τους υπόλοιπους. Την περασμένη φορά η απόφαση του Προέδρου ήταν ότι δεν θα έπρεπε να είναι γνωστές, ε, γνωστοί ποιοι έχουν υπογράψει. Αποφασίσαμε όμως ε, ομοφόνος αυτή τη φορά ότι για λόγους διαφάνειας οι υπογραφές αυτές πρέπει να είναι δημόσιες, να ε, δημοσιεύονται γιατί εμείς κηρύσουμε την διαφάνεια και πρέπει πρώτα εμείς να είμαστε διαφανείς. Μετά μιλήσαμε για τις ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων. Η Επιτροπή μας θα είναι παρούσα την ακρόαση 7 Οκτωβρίου του ε, υποψήφιου Επιτρόπου Τίμερμανς και επίσης μας, έχει, μας έχουν προσκαλέσει στην ακρόαση του κυρίου Ναυράτσκι, η Επιτροπή Πολιτισμού μας κάλεσε και επειδή η αρμοδιότητά μας ε, είναι η πρωτοβουλία των ε, πολιτών και επειδή είμαστε πολύ κοντά στους πολίτες γιατί είμαστε ε, η μοναδική επιτροπή που είναι τόσο κοντά στους πολίτες και επειδή ο κύριος Ναμπράσκη θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του πολιτισμού υπάρχουν πολλά, πολλοί τομείς που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. Οπότε ελπίζω να σας δω στις ακροάσεις αυτές. Ε, η Επιτροπή του ε, Κοινοβουλίου της Σκοτίας ε, θα έρθει στις, στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίναμε επίσης τις δραστηριότητες το 2015 και ζητούμε επίσης και νομική γνωμοδότηση για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας πολωνό δικηγόρο και επίσης ζητήσαμε, μιλάμε για τη διερευνητική επίσκεψη που έγινε στη ΣΥΑ το 2014 ε, Πρόκειται για μια παραβίαση πνευματικής, δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και πρέπει να εξετάσουμε την αποστολή ε, στον αναφέρονται για το θέμα αυτό. Μπορούμε να εγκρίνουμε τα συμπεράσματα των συντονιστών. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της 7ης Οκτωβρίου, έχει διανεμηθεί. Εγκρίθηκε από τους συντονιστές, σας το λέω απλώς ενημερωτικά. Υπάρχουν ερωτήσεις? Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με τις ε, αποστολές μας, ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά, το γνωρίζουμε αυτό, έχουμε καθυστερήσει και λίγο. όλα αυτά, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητο και επίγον να γίνει μια αξιολόγηση όπως ζητήθηκε άλλωστε ομοφόνος από την ομάδα των σοσιαλιστών να οργανωθεί το συντομότερο δυνατόν μια αποστολή στη Λαμπεντούζα. Χωρίς καθυστέρηση, να μην περιμένουμε δηλαδή τους πρώτους μήνες του 2015, δεν πρόκειται για μια αποστολή ρουτίνας ούτε μια, για μια απλή επίσκεψη, και δεν θα έλεγα ότι είναι απλώς μια διερευνητική επίσκεψη. Στη Μεσόγειο λαμβάνουν καθημερινά χώρα ε, δραματικά γεγονότα και κυρίως ε, πρόκειται για ένα μήνυμα αλληλεγγύης η οποία την οφείλουμε και για την αναγνώριση αυτών των γεγονότων κυρίως μετά από το όσα είπε το Συμβούλιο της Ευρώπης που εντόνως ε, μίλησε για το θέμα ότι πραγματικά δεν γίνεται τίποτα στην ουσία για να αποφευχθεί το εμπόριο ανθρωπίνων ε, ανθρώπων. Και γι' αυτό και θα ήθελα και πάλι να επιστήσω την προσοχή σας ότι στο γεγονός ότι είναι σκόπιμο να αξιολογήσουμε λειτουργήσουμε με προσοχή και με ευαισθησία ε, που όλοι έχουμε τη, τη δυνατότητα να πάμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και ακριβώς επειδή τις επόμενες ημέρες ε, θα είναι η επέτειος της ε, λυπηρότατης καταστροφής της Λαμπεντούζα στις 3 Οκτωβρίου που κόστησε τη ζωή σε 303 άτομα. Το θέμα αυτό δεν έχει ακόμα λυθεί και θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα και θα ήθελα να ζητήσω και από τους συναδέλφους να στηρίξουν αυτή την πρότασή μου. Η κυρία Βαλίνα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς απλά και μόνο ένα σχόλιο για την ημερήσια διάταξη, για το θεματολόγιο λυπούμαστε που ε, δεν, έχει, δεν βρίσκεται για σήμερα το θέμα των πετρελαϊκών ερευνών, αλλά χαιρόμαστε για το ότι για τις 7 Οκτωβρίου το έχει προβλέψει και το έχει συμπεριλάβει η Πρόεδρος ε, στην ημερήσια διάταξη. Επήγει το θέμα αυτό, διότι οι πετρελαϊκές έρευνες που προβλέπεται να αρχίσουν τον Νοέμβριο, κάνουμε λόγο για ένα πολύ, μια ιδιαίτερη περιοχή κοινοτικού ενδιαφέροντος και συμφέροντος, ε, στα Κανάρια νησιά δηλαδή, στο κέντρο ακριβώς του κοινοτικού αυτού συμφέροντος και ενδιαφέροντος. Και ελπίζουμε ότι στις 7 Οκτωβρίου θα τηρηθεί η υπόσχεση της Προέδρου και δεν θα αναιρεθεί και θα εξεταστεί το θέμα αυτό. Κύριος Χατζηγεωργίου παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ε, νομίζω ότι είναι καλά να δημιουργηθεί μια πλειοψηφία εδώ που να βάρει το βάρος της υπέρ της άποψης που ελέγχθη προηγουμένως για επίσκεψη ομάδας ερεύνησης στη Λαμπετούσα. Και νομίζω ότι πρέπει να, να μην μείνουμε πάνω στην απόφαση ότι αυτές οι επισκέψεις μπορούν να γίνουν μόνο μέσα στο 2015. Ε, έχει αναλυθεί επαρκώς, έχουν αναλυθεί επαρκώς οι λόγοι ε, από την συνάδελφο και νομίζω πως αν και άλλοι συνάδελφοι δημιουργήσουμε εδώ μια πλειοψηφούσα άποψη ότι πρέπει να γίνει μια επίσκεψη στη Λαμπετούσα να το κάνουμε. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία είναι ανάγκη να γίνει επίσκεψη πριν το 2015, όπως είναι το θέμα της αμοχώστου που υπάρχει ήδη αναφορά ενώπιον μας. Όμως ε, για αυτό το θέμα θα το κρατήσω για το 2015, θα σας στείλω σήμερα επιστολή που θα ζητά να υπάρξει ε, fact-finding mission ε, και για την αμόχωστού Όμως ε, το θέμα της Λαμπεντούσα νομίζω ότι είναι καλό εδώ να φανεί αν υπάρχει μια πλειοψηφία που λέει αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ. Monsieur Martin, s'il vous plaît. Oui, merci. Simplement, moi, je... Ευχαριστώ. Και εγώ υποστηρίζω μια επίγουσα αποστολή στη Λαμπεντούζα. Συμφωνώ με αυτό. Νομίζω ότι ε, ο ίδιος ο πρόεδρος του Μάρτιν, ο Μάρτιν Σούλτς αλλά και πολλοί άλλοι είχαν ζητήσει κάτι τέτοιο. Το θέμα της Λαμπετούζα είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορούμε να στείλουμε το μήνυμα ότι καθυστερούμε ή ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά για να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα ενώ υπάρχει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση σε, αυτό, σε αυτή την πόλη ε, που πλήττεται σήμερα από μαζική άφηξη μεταναστών οπότε νομίζω ότι πρέπει επιγόντως να μετα μεταβούμε στη Λαμπεντούζα. Οπότε συμφωνώ με την ιδέα αυτή. Κύριε Μάρια. Κύριος Μαριάς παρακαλώ. Είχαμε επισημάνει και άλλη φορά ότι οι επισκέψεις στα κράτη-μέλη ε, για fact-finding missions πρέπει να γίνουν άμεσα και για τον λόγο αυτό είχαμε διαφωνήσει με την άποψη που επικρατούσε ότι δεν υπάρχουν πόροι, δεν υπάρχουν χρήματα για να γίνουν αυτές οι δραστηριότητες το 2014. Και το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Βεβαίως αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός για το 2015. Όμως η πρόταση που θέτει η συνάδελφος είναι πάρα πολύ επίγουσα και γιατί στη Λαμπεντούζα υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και γιατί αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές και επίσης οι αφήξεις ε, από χώρες όπως είναι, ε, ο Λίβανο, ε, όπως είναι η Συρία, όπως είναι η Λιβύη λόγω και των πολεμικών συγκρούσεων που υπάρχουν στις περιοχές αυτές και αυτή η πίεση προσφύγων προς την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεράστια. Αφορά βεβαίως και την Ελλάδα, όπου και εκεί έχουμε μια τεράστια πίεση. Νομίζουμε λοιπόν ότι στο βαθμό που υπάρχει δυνατότητα θα πρέπει να πάμε στη Λαμπεντούζα για να στείλουμε και ένα μήνυμα ότι η Επιτροπή Αναφορών και το Κοινοβούλιο παρακολουθεί τα ζητήματα αυτά ούτως ώστε να είμαστε κοντά στους πολίτες και ταυτόχρονα να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει για να μπορέσουμε να επιμείνουμε, να πιέσουμε να ληφθούν σοβαρά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πιέσεις, με τις αφήξεις τεραστίου αριθμών προσφύγων αλλά και άλλων μεταναστευτικών ροών. Ευχαριστώ. Κάνω την εξή πρόταση ίσως. Πρώτον, και εγώ αναγνωρίζω πρέπει να πω τα προβλήματα που επικρατούν στην Λαμπεντούζα. Δεύτερο, μέσω της Προέδρου θα ήθελα να παρακαλέσω αυτή την κατάσταση να την συνεξετάσουμε στην διάσκεψη των Προέδρων. Διότι αυτό το οποίο αναφέρθηκε σωστά πιο πριν, αυτό είναι η υπόθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Πρέπει να συντονιστούμε δεν είναι δυνατόν κάθε εβδομάδα μια νέα κοινοβουλευτική επιτροπή να αναφύεται και να αναδύεται στην Λαμπεντούζα. Πρέπει να συντονίσουμε το έργο μας από πλευράς Ευρωβουλής. Θα προτιμούσα, Πρόεδρε, και αυτό να ψηφιστεί στην, προ... στην διάσκεψη των Προέδρων προς έγκριση. Ίσως υπάρχουν και άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές που σχεδίαζαν κάτι ή όχι, αλλά πρέπει να είναι συντονισμένη η δράση μας. Και τρίτον, οι συντονιστές δεν ήταν αρνητικοί ή κακοί επειδή είπαν δεν θα γίνει fact-finding mission πλέον πρέπει να πούμε έχουμε τεράστιο αριθμό 2.000 αναφορών που έχουμε ακόμα στις αποσκευές μας ε, από το παρελθόν. Πρέπει να δούμε σε σχέση με τους αναφερόμενους που εδώ και χρόνια δεν έχουν τύχει απάντησης επειδή δεν ολοκληρώθηκε η εξέταση της αναφοράς τους, είπαμε θα κάνουμε πρώτα τη δουλειά μας, τα καθήκοντά μας. Εκείνοι που κατεπηγόντως θέλουν να αποχωρήσουν, ζητώ κατεπηγόντως να βοηθήσουν, να συνεισφέρουν, να καλύψουμε τις υποχρεώσεις του παρελθόντος. Και τότε μπορούμε να δούμε προτάσεις για fact-finding missions για το μέλλον και πού μπορούμε να πάμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτά η διάσκεψη των Προέδρων, από κοινού και με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, θα πρέπει μια συντονισμένη διαδικασία να υιοθετήσουμε. Ελένη, σε παρακαλώ. Η Ελένη Θεοχάρους, παρακαλώ. εγώ θα συμφωνούσα με τον συντονιστή ότι είναι πολλά τα σημεία στα οποία θα ε, μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε επίσκεψη για fact-finding mission, ε, δεδομένου ότι είναι πολλά τα, τα ζέοντα, τα, θερμά σημεία στην Μεσόγειο. Για παράδειγμα είναι η Σάμος, ε, είναι άλλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είναι η ίδια εκεί προσωπού έχουμε τεράστια ροή προσφύγων από τη Συρία στα κατεχόμενα και από εκεί διοχετεύονται παράνομα στις ελεύθερες περιοχές. Πρόσφατα ξύλωσε η Κυπριακή Αστυνομία ένα τεράστιο ε, δίκτυο και μάλιστα τζιχαντιστών. Ήταν, υπήρχε αναφορά στις εφημερίδες. Η Λαμπεντούζα είναι μια σοβαρή περίπτωση την οποία πρέπει να ειδούμε. Αλλά παράλληλα πρέπει να σκεφτούμε ότι και η Μάλτα δέχεται την ίδια πίεση. Άρα θα πρέπει να κάνουμε κάποιου συνδυασμού, ώστε όλα τα ε, φλέγοντα σημεία της νότιας ε, της ε, Μεσογείου να τα δούμε συγκεντρωμένα. Μια αποστολή στη Λαμπεντούζα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα ήταν απλώς μια αποσπασματική εκτίμηση του προβλήματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Okay. Let me try to conclude. Μάλιστα, να προσπαθήσω να συνοψίσω. Καταρχάς, λάβαμε στους συντονιστές μια ομόφωνη απόφαση τον Ιούλιο να μην γίνουν τέτοιου είδους αποστολές διερευνητικές ε, κατά τη διάρκεια του 2014. Ήταν ομόφωνη απόφαση, κανένας δεν διαφώνησε τότε. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι πρέπει να πάρουμε σοβαρά αυτά που συμβαίνουν στη Λαμπεντούζα και ε, σε άλλα μέρη της Μεσογείου, ε, σε παράκτιες περιοχές και σε νησιά. Εμείς ε, είχαμε επισήμως στείλει μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ πριν από δύο χρόνια και είχαμε ζητήσει να μας στείλουν την έκθεση που προέκυψε γιατί η αντιπροσωπεία πήγε και στη Λαμπεντούσα και στη Σικελία. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επανεφευρίσκουμε τον τροχό κάθε φορά έχει γίνει ε, δουλειά από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς αυτή την κατεύθυνση και υπάρχουν συμπεράσματα από, τη συγκεκριμένη αντιπροσωπεία, αλλά μπορούμε να καλέσουμε στην επόμενη μας συνεδρίαση την Ιταλική Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι να λάβουν αυτήν την ενημέρωση από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για να έχουμε μία εις βάθος συζήτηση για το θέμα αυτό. Να καλέσουμε και τους ε, ε, αναφέροντες και να συζητήσουμε και το θέμα αυτό της Λαμπεντούζα. Είναι ίσως πιο αποτελεσματικό αυτό από το να πάμε εκεί. Γιατί όπως είπε και ο κύριος Γιάρ ήδη, υπήρξαν πολλές αντιπροσωπείες κρατών μελών που πήγαν στην, στο νησί και τίποτε δεν έγινε. Οπότε πρέπει να ε, το λάβουμε και αυτό σοβαρά υπόψη, εν ώψη των ακροάσεων με τους υποψήφιους επιτροπούς, τι έχει σκοπό να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην περίπτωση αυτή που ε, πρόσφυγες πεθαίνουν ε, είτε στη Λαμπεντούζα είτε στη Μεσόγειο, σε άλλα μέρη της Μεσογείου. Τεράστιες τραγωδίες λαμβάνουν χώρα κάθε μέρα μόνο το Σεπτέμβριο πάνω από 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μεσόγειο προσπαθώντας ε, να ζητήσουν διεθνή προστασία στην Ευρώπη. Αυτό είναι τραγωδία και πρέπει οπωσδήποτε κάτι να κάνουμε. Γιατί λοιπόν να μην αποφασίσουμε μαζί ότι στην επόμενη συνεδρίασή μας θα έχουμε μία εμπεριστατωμένη συζήτηση με τους αναφέροντες, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδεχομένως να καλέσουμε και την Ιταλική Προεδρία. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας από αυτού. Τάκη. παρακαλώ. Να πω ότι τα καταληκτικά σας σχόλια νομίζω ότι πράγματι δίνουν μια σωστή λύση και μια καλή διέξοδο. Άλλωστε είμαστε στο Σεπτέμβριο, το 2015 δεν είναι μακριά. Ε, όμως θέλω να πω ότι η αναφορά πως υπήρξε απόφαση στους coordinators ε, δεν πρέπει να αποτελεί μια τελική απόφαση. Εδώ πρέπει να παίρνονται αποφάσεις. Οι coordinators δικαίωμά του σωστό να σκεφτούν και να δώσουν καθοδήγηση. Αλλά δεν μπορεί να αποτελεί την τελική απόφαση η απόφαση των coordinators. Όμως επαναλαμβάνω τα καταληκτικά σας σχόλια νομίζω ότι δίνουν λύση στο πρόβλημα. May I just ask you, do you, do you mean, do you mean that you want Θέλετε λοιπόν να ξανανοίξουμε τη συζήτηση αυτό εννοείται και να πάρουμε μια νέα απόφαση ή να παραμείνουμε στην απόφαση που ομοφόνους είχαν λάβει οι συντονιστές. Να μείνουμε πάνω στην απόφαση που έχουν μέσα τα καταληκτικά σας σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. sorry, the, the, Τα γυαλιά μου, τα ακουστικά μου, το μικρόφωνο, περδεύτηκα κάπως. Εντάξει, τα κατάφερα όμως. Είναι εδώ ο ε, διευθυντής ε, Πασκάλ Νεαρντίνη, ο οποίος θα μας πει ορισμένα πράγματα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη συνεργασία της με την Επιτροπή Αναφορών και μετά την παρουσίασή του θα γίνουν ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ευκαιρία η αρχή της νέας κοινοβουλευτικής θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας να κάνουμε μια πολύ καλή συζήτηση για την συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιτροπής Αναφορών. Όπως γνωρίζετε η Επιτροπή βρίσκεται επίσης σε μεταβατικό στάδιο, θα έχουμε μια νέα ομάδα σε μερικές εβδομάδες, οπότε όλο και περισσότερο δικαιολογείται αυτή η συζήτηση με την Επιτροπή Αναφορών ε, δεν χρειάζεται να σας πω ότι είναι η αναφορά βάσει των συνθήκων ένα δημοκρατικό εργαλείο, πολύ σημαντικό και κατά τη διάρκεια των ετών υπήρξε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Αναφορών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει μια σημαντική αύξηση στον αριθμό των αναφορών και βεβαίως συνεπώς και στο φόρτο εργασίας ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που πρέπει να απαντήσει στις αναφορές αυτές και στα λίγα λεπτά που μου έχετε δώσει θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω κάποια προβλήματα, κάποια ζητήματα που παραμένουν έκρεμοι και ε, τον τρόπο με τον οποίο πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα έπρεπε να καλυφθούν τα ζητήματα αυτά. Καταρχάς, ε, να δούμε κάποια αριθμητικά στοιχεία. Έχου, έχει λάβει η Επιτροπή Αναφορών το 2013 πολύ μεγαλύτερο αριθμό αναφορών, 45% αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και πολλές από αυτές τις αναφορές πράγματι καταλήγουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 45% όλων αυτών των αναφορών ε, αφορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι το 60% όλων των παραδεκτών αναφορών. Σε απόλυτους όρους αυτό σημαίνει 1.250 περίπου αναφορές το 2013 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τομείς ε, ε, που πραγματεύονται οι αναφορές, προστασία περιβάλλοντος, απόβλητα, ύδατα, ε, ποιότητα των υδάτων, ε, αξιολόγηση επιπτώσεων πριν ε, από μεγάλα ε, πριν από μεγάλες δημόσιες προμήθειες, ε, θεμελιώδη δικαιώματα όπως η οικογενειακή επανένωση, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ε, μειονότητες, αναπηρίες, τρίτον, ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, των εργαζομένων, αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων και τέταρτος τομέας, οικονομική και κοινωνική κρίση, υπήρξαν πολλές αναφορές ε, για θέματα τραπεζικά, στέγασης κλπ. Ένας μικρός αριθμός υπηρεσιών λοιπόν, όπως η Γενική Διεύθυνση, ΜΑΡΚΤ, ε, ε, περιβάλλοντος και σε μικρότερο βαθμό οικονομικών πρέπει να, να, απαντήσουν στις αναφορές αυτός αναφορές αυτές. Προσπαθούμε εντός τριών μηνών να δώσουμε απάντηση. Αυτή είναι μια ε, συμφωνία που έχουμε με την Επιτροπή σας. Κάτι το οποίο βέβαια είναι πολύ απαιτητικό ως προθεσμία γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη και όλες τις ε, μεταφραστικές ανάγκες και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ζητήσει και πληροφορίες για από τα κράτη-μέλη ε, και από τις διάφορες αρμόδιες αρχές. Υπάρχει μόνο η Γενική Γραμματεία ως σημείο εισόδου μετά γίνεται ανάθεση σε, κάποια, σε μια από την αρμόδια, σε μια αρμόδια επιτροπή, ε, σε καμιά αρμόδια υπηρεσία ή σε συναφείς υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, υπάρχει τελικά μια ανακοίνωση που είναι ο τρόπος με τον οποίο απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνεται από την Γενική Γραμματεία ώστε να εξασφαλιστεί έλεγχος ποιότητας αλλά και ότι η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει μπορέσει να γνωμοδοτήσει. Ε, μετά υποβάλλουμε τα έγγραφα αυτά, τις ανακοινώσεις, σε παρτίδες κάθε μήνα. Ε, στέλνουμε εκατοντάδες ε, ανακοινώσεων που απαντούν στις αναφορές. 741 ανακοινώσεις στείλαμε το 2013 και στους 8 πρώτους μήνες αυτού του έτους έχουμε ήδη φτάσει τις 806 ανακοινώσεις. Οπότε βλέπετε πόση πίεση υπάρχει. Φυσικά είναι ευνόητο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παρούσα στις συνεδριάσεις σας και μας δίνεται και το λόγο να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και να δώσουμε λεπτομέρειες στον τρόπο απάντησης στους αναφέροντες. Κάτι το οποίο έχουμε επίσης δει πολλές φορές είναι ότι υπάρχουν πολλές φορές επιπρόσθετες ανάγκες για περαιτέρω διευκρινήσεις μετά από την πρώτη εξέταση. Πολλές φορές χρειάζεται να ξαναέρθουμε σε επαφή σε περίπτωση διαδικασίας παραβάσεων κατά κρατών μελών. Πρέπει να περιμένουμε τις απαντήσεις των των εθνικών αρχών και αυτό βέβαια σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει μεν ε, αυστηρή ε, προθεσμία, ε, όμως υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, ανταλλαγή στοιχείων και μερικές φορές χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν όλα αυτά. Φτάνω τώρα στο σημαντικό σημείο της παρουσίασής μου, ποια είναι τα βασικά ε, προβλήματα. Κάποιοι από εσά έχετε ήδη αναφέρει ότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, αναφορές, πάνω από 2.000 που εκκρεμούν. Ε, εμείς ευχαρίστως να προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε και να δίνουμε όσο το δυνατόν, μια, όσο δυνατόν συντομότερα μια απάντηση στους πολίτες. Πιστεύουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει με το θέμα του παραδεκτού των αναφορών ε, τη στιγμή που λαμβάνονται οι αναφορές ε, γιατί εσείς ε, και οι συνάδελφοί σας στη Γραμματεία αλλά και εμείς στην Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρειάζεται να εξετάσουμε το παραδεκτό χαρακτήρα ε, και τελικά καταλήγουμε ότι δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν βρούμε έναν, λοιπόν, ένα μηχανισμό λοιπόν μέσω του οποίου θα μπορέσουμε πράγματα τα οποία ε, δεν απευθύνονται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράδειγμα κακοδιαχείριση ε, για την οποία κατηγορείται κάποιο ευρωπαϊκό όργανο ε, ο, Ευρωπαϊ... ο Ευρωπαίος μπορεί επίσης να αναλάβει δράση και αυτό θα απλοποιούσε τα πράγματα όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών μελών. Δεύτερο σημείο. Ξέρετε ότι δεν μεταγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τα κράτη-μέλη τις οδηγίες. Και σε μερικά κράτη-μέλη αυτό σημαίνει διάφορα επίπεδα ε, διαχείρισης, ε, τοπική αυτοδιοίκηση, περιφερειακή αυτοδιοίκηση και πιστεύουμε ότι σε μερικές περιπτώσεις θα ήταν πολύ χρήσιμο τα κράτη-μέλη να καλούνται στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών και να παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται κάποιο συγκεκριμένο νομοθέτημα. Είμαστε ευγνώμων στον προκάτοχό σας γιατί προσπάθησε να ομαδοποιήσει τις ε, αναφορές ε, σε τομείς, ε, κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία στην Επιτροπή. Έχουμε όμως ένα τεράστιο ρυθμό εκρεμών αναφορών που παραμένουν εκρεμίσει για πολλά χρόνια και μερικές μάλιστα δεν παρουσιάζουν και ιδιαίτερη εξέλιξη είτε επειδή υπάρχει διαδικασία ε, παράβαση, είτε επειδή περιμένουμε τα αποτελέσματα μιας νομοθεσία που καλύπτει το θέμα αυτό. Και πρέπει να παρακολουθούμε, πρέπει να διαχειριζόμαστε όλες αυτές τις ε, αναφορές και ενδεχομένως να πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο κατηγοριοποίησης ε, όλων αυτών των αναφορών. Οι προτάσεις τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπα το θέμα του παραδεκτού ε, χαρακτήρα, τη στιγμή που λαμβάνεται η αναφορά, για να μπορούμε να στρέφουμε τους αναφέροντες ε, προς τη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά τώρα τις ε, εκρεμείς αναφορές και μιλάω για την έκθεση Βαλένσα, όπου αναφέρεται ότι κάποιες αναφορές παραμένουν εκρεμείς χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι. Μία ιδέα θα ήταν ίσως ότι κάποιες από αυτές τις αναφορές ε, για τις οποίες υπάρχει ανοιχτή διαδικασία επί παραβάση, τουλάχιστον να υπάρχει κάποιο είδους επισήμανση ε, ως ε, ιδιαίτερη περίπτωση όταν υπάρχει μια διαδικασία επί παραβάση ανοιχτή, οπότε να μπορούμε να τις βάλουμε σε μία ομάδα και να επανέλθουμε σε αυτές. αφή στιγμής στιγμή η διαδικασία επιπαραβάση έχει περάσει σε δεύτερο ή τρίτο στάδιο. Δηλαδή υπάρχει μία σχέση στον τρόπο με τον οποίο ε, μπορεί να συνεχίσουν ε, οι αναφορές ε, να εξελίσσονται και η ε, και στη συνέχιση της διαδικασίας επί παραβάση. Επίσης έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι πρέπει να ανταποκρινόμαστε γρήγορα στις αναφορές. Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα με μονομένα εφαρμογής. Δεν μιλάω για ένα γενικό ε, πρόβλημα κακής εφαρμογής ή για μαζικά προβλήματα τα οποία ε, θα χρειάζονταν άλλου είδους μέσα. Μιλάω για έναν άνθρωπο που έχει ένα δίπλωμα που δεν μπορεί να αναγνωριστεί σε ένα άλλο κρατος μέλος ή ένα άτομο το οποίο εισάγει μία χώρα από μία, ε, από μία χώρα και δεν μπορεί να το ε, καταχωρήσει στην άλλη χώρα. Έχουμε το Solvit που είναι ένας ε, μηχανισμός στο διαδίκτυο που μπορεί να βοηθήσει την επίλυση τέτοιου είδους διαφορών Ίσως θα μπορούσαμε λοιπόν να διαφημίσουμε λίγο περισσότερο τέτοιου είδους ε, μηχανισμούς. Το θέμα της συμμετοχής των κρατών μελών το ανέφερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Αν τα κράτη-μέλη δεν συμμετέχουν στη συζήτηση αυτή στην Επιτροπή Αναφορών, εμείς πρέπει να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, δεν έχουν ακούσει ακριβώς ε, πώς έχουν οι αναφορές και χάνουμε πάρα πολύ χρόνο βεβαίως. Και τέλος, θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας με την Επιτροπή σας. Έχουμε πει ότι θα μπορούσαμε με τη Γραμματεία να έχουμε προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις πριν από τις ε, τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής σας, να εξετάζουμε την ημερήσια διάταξη, να είμαστε βέβαιοι ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι είναι παρόντες στις συζητήσεις. Και ολοκληρώνοντας, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και πάλι να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απολύτως έτοιμη να συνεργαστεί μαζί σας για να μπορεί μπορέσουμε να ευθυγραμμίσουμε κάπως τις διαδικασίες ε, και να επιταχύνουμε ε, την εξέλιξη των αναφορών ε, με σκοπό την ικανοποίηση των πολιτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λεαρντίνη. Τώρα να ακούσουμε ερωτήσεις. Margaret κυρία A Έχω μπερδευτεί λιγάκι λέτε να κλείνουμε κάποιες αναφορές ε, χωρίς ε, να συμμετέχουμε εμεί. Αν υπάρχει μια διαδικασία επί παραβάση, τότε δεν υπάρχει λόγος να κλείσουμε την αναφορά. Για παράδειγμα υπάρχουν αναφορές που παραμένουν ανοιχτέ και επανέρχεται το ίδιο θέμα το οποίο πραγματεύεται η αναφορά συνεχώς. Το 2009, ας πούμε, υπήρχε μια τέτοια ή τέτοιου τους αναφορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να κάνει οτιδήποτε, κάτι το οποίο ήταν θλιβερό γιατί αφορούσε πάρα πολλούς πολίτες. Εξακολουθούμε για το ίδιο θέμα να λαμβάνουμε πολλές αναφορές. Εντάξει, η Ισπανική κυβέρνηση λέει ναι, απαντήσαμε στο αίτημά σας κλπ. Αλλά συνεχίζονται οι εξελίξεις. Και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. τα θέματα, ας πούμε, της επεξεργασίας αποβλήτων. Και μας είπατε ότι ίσως θα έπρεπε περισσότερο τα κράτη-μέλη να είναι παρόντα. Ένα από τα βασικά προβλήματα στην Ιταλία ήταν ότι κανένας δεν ήταν υπεύθυνο. Κάναμε συζητήσεις με την Ιταλική κυβέρνηση και ο ένας πετούσε τον παλάκι στον άλλον. Κανένας δεν αναλάμβανε την ευθύνη για το πρόβλημα που συζητούσαμε. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να το διαχειριστούμε αυτό στο μέλλον, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία της Ένωσης εφαρμόζεται σωστά στις χώρες, ακόμη και όταν υπάρχει αυτό το διοικητικό χάος. Ε, μπορώ να σας πω, ας πούμε, ότι πήγαμε στην Καμπανία και εκεί ο Υπουργός μας είπε ότι έπρεπε να συμφωνήσει με 561, 561 δημάρχους για να προχωρήσει το θέμα που συζητούσαμε. Πείτε μας λοιπόν, πώς πιστεύετε ότι πρέπει να διαχειριστούμε κάτι τέτοιο, που πραγματικά είναι πολύ δύσκολο για μας. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα περιορίσω όλους τους άλλους ομιλητές στο ένα λεπτό, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε στην ημερήσια διάταξη. Και θα έρθει και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητή τη 11.30 και πρέπει να κλείσουμε κάποιε αναφορέ μέχρι τότε. Βίκτορ, ξέρει. Πρέπει λοιπόν να είστε πολύ σύντομοι. Ναι, ευχαριστώ και άλλη μια φορά ρητά. Παράκλησή μου απλά είναι η Επιτροπή τις προτάσεις από κοινού με εμάς να τις συζητήσει και να τις αναλύσει. Έχουμε και αυτό το διοικητικό έγγραφο και έχουμε πολλά πράγματα που επαναλαμβάνονται. Η ανάλυση επί των προβλημάτων είναι η ίδια και όταν βλέπουμε 60% των αναφορών περνούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τότε το υπόλοιπο 40% τι είναι. Είναι πάρα πολλές μη παραδεκτές και άλλες. Ε, χρειάζεται λοιπόν ένα φίλτρο διήθησης και το θέμα του παραδεκτού, αποδεκτού ή όχι και της ε, αρμοδιότητας, ε, admissibility και responsibility θα πρέπει να βρούμε το δυνατόν γοργότερα τον διαβλό, τον τρόπο να συνεχίζεται, να τύχει συνέχεια μια, ε, μια αναφορά ή όχι. Με τον Ombudsman το ίδιο πρόβλημα θα δούμε ότι έχουμε σε σχέση με ε, θέματα αναφορών. Παράκλησή μου, σύντομα, πολύ απλά. Θα πρέπει λοιπόν από το έγγραφο αυτό να δούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι τα προβλήματα και πού έγκυνται. Είναι σχεδόν τα ίδια. Χρειάζεται ένα φίλτρο διήθησης για να δούμε τι θα γίνεται με την αποδεκτότητα, παραδεκτότητα και να επιλύονται τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Thank you. Soledad, Ευχαριστώ, παρακαλώ. Εγώ θέλω να πω ότι πρώτον αυτό που φαίνεται με μια πρώτη ματιά ότι είναι ένα πρόβλημα είναι μια καλή είδηση. Καλά μαντάτα για τους ε, πολίτες που αισθάνονται απογοήτευση σε σχέση με τα θεσμικά όργανα. Και έχουμε και μια σημαντική αύξηση λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Αυτό είναι θετικό. Πρέπει να βρούμε μια μέθοδο μεθοδολογικά για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα και να είμαστε επαρκείς ε, και εναντί της Επιτροπής. Πρέπει οι αναγκαίοι πόροι να διασφαλίζονται ώστε να μπορούμε να τα επιλύουμε για την παραδεκτότητα, την το αποδεκτό ή όχι και φυσικά έχει δικαίωμα ο αναφέρον να απευθύνεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Σε σχέση με τις αρμοδιότητες πρέπει να δούμε πώς θα επιληθεί το πρόβλημα να ενημερώσουμε τον πολίτη άμεσα και μέσω της ιστοσελίδας ποιος είναι ο ρόλος ο δικός μας που μπορούμε να διασφαλίσουμε και πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε να επιληθεί το πρόβλημα αρμοδιοτήτων. Αυτό είναι ένα πρώτο. Και μετά στη συνέχεια είναι αναγκαίο πραγματικά να βρούμε τον τρόπο να βρούμε τι γίνεται σε σχέση με την αρμοδιότητα και τις ευθύνες από πλευράς των μελών μας, ώστε να υπάρχει το δυνατόν μικρότερη ανάμιξη σε σχέση με την αντιμετώπιση των αναφερών από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί, διότι πολλές φορές βλέπουμε σε σχέση με ε, τους όσους κυβερνούν, τις κυβερνήσεις, πολλές φορές ότι υπερβαίνουν τα εσκαμμένα και πρέπει πραγματικά με τους πολίτες, ε, με το δικαίωμα αναφοράς που έχουν να είμαστε διάφανοι, να διασφαλίζεται η διαφάνεια σε σχέση με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Mr. Κύριος Μαριάς παρακαλώ όπως έχουμε επισημάνει και άλλες φορές, το δικαίωμα αναφοράς είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως αυτό πρέπει να ασκείται και ταυτόχρονα εμείς ως Επιτροπή πρέπει να μπορούμε να ανταποκριθούμε στην ενάσκηση αυτού του δικαιώματος. Βεβαίως υπάρχουν ε, αναφορές οι οποίες δεν είναι παραδεκτές και αυτές θα απορρίπτονται. Αλλά δεν μπορούμε να σταθούμε σε μια στενή ερμηνεία του παραδεκτού ούτως ώστε να ξεπετάξουμε διάφορες αναφορές επειδή υπάρχει μεγάλος αριθμός αναφορών. Δεύτερο, ε, μου έδωσε την εντύπωση η Επιτροπή ότι ε, θέλει λίγο να ξεφορτωθεί τις αναφορές οι οποίες είναι πάρα πολλές. Θα πρέπει να αντιληφθεί ότι και η Επιτροπή και εμείς ε, επιτελούμε ένα σημαντικό ρόλο και το ότι απευθυνόμαστε στην Επιτροπή αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας των θεσμικών οργάνων και αν θέλετε τις δίνουμε μια μεγαλύτερη ευκαιρία και τις δίνουμε και ένα feedback για το πώς εφαρμόζεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διάφορα κράτη-μέλη. Προκειμένου εν συνεχεία η Επιτροπή να ασκήσει και τα δικά της αυτοτελή δικαιώματα που είναι ο έλεγχος των κρατών μελών σε σχέση με την πραγματική, την ορθή εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως εδώ πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία των δύο θεσμικών οργάνων και ταυτόχρονα μια αποφασιστικότητα απέναντι σε, στα κράτη-μέλη, σε όλα τα επίπεδα, είτε στο επίπεδο κυβερνήσεων είτε στο επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να υπάρξει η πραγματική εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η τήρηση των δικαιωμάτων των πολιτών. Άρα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να κινηθούμε και να είμαστε αποτελεσματικοί και να μην έχουμε διάφορες αναφορές που πηγαίνουν και έρχονται μεταξύ της δικιάς μας Επιτροπής και της Κομισιόν και δεν βρίσκουμε άκρη. Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα ζητήματα και να ελέγχονται. Το τι απαντά ένα κράτος μέλος ότι δήθεν τηρεί τις διαδικασίες του κοινοτικού δικαίου δεν σημαίνει ότι είναι και ορθό ή ότι είναι και αληθές. Πρέπει αυτά να ερευνώνται ούτως ώστε να παίρνουμε αποφάσεις που να βοηθούν πραγματικά στην ενάσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Ε, κυρία Θεοχάρου, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο ρόλος της Επιτροπής νομίζω ότι είναι η ε, υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, η προστασία τους από την αυθαιρεσία της εξουσίας και δυστυχώς έχουμε αυθαίρετες εξουσίες σε όλη την Ευρώπη αλλά και η ανάδειξη του ρόλου του καλού Ευρωπαίου πολίτη. Γι' αυτό, κυρία Πρόεδρε, δεν ξέρω αν ισχύει ένας τέτοιος θεσμός, αλλά η δική μου πρόταση θα ήταν αν κάποιες από τις ε, αναφορές στην Επιτροπή μας κρίνονται ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ή ότι ε, έχουν ένα ιδιάζον στοιχείο, να ανοίγουμε ένα δημόσιο διάλογο online για κάποιο χρονικό διάστημα που να δίνουμε την ευκαιρία σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες πρώτον να καταθέτουν τις δικές τους τις θέσεις για την συγκεκριμένη αναφορά και δεύτερον να αν έχουν ανάλογα προβλήματα σε άλλα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας γνωστοποιούνται ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα το οποίο θα βγαίνει από την αναφορά αυτά να αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να καλύπτει πολλές ε, ανάλογες περιπτώσεις και ενδεχομένως να μειώσουμε και τον μεγάλο αριθμό των ε, αναφορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Και τώρα έχω την Πεατρίση στον κατάλογο. Να κλείσουμε μετά τον κατάλογο, γιατί πρέπει να ξαναδώσουμε το λόγο στην ε, Επιτροπή και να προχωρήσουμε. Συμφωνεί. Ωραία. Πεατρίση, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο της Επιτροπής για την παρουσίασή του και τα στοιχεία που μας έδωσε. Είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε ότι με αύξηση στον αριθμό των αναφορών δεν είναι αναγκαστικά ένα θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση των εργασιών μας υπό εξέλιξη. Με άλλα λόγια, όπως είπε η συνάδελφος Άουκεν πιο πριν, είναι σημαντικά τα όσα λέγονται και τα ονόματα και περισσότερες αναφορές δεν είναι υποχρεωτικά ο καλύτερος ορισμός για το τι μπορεί να γίνει από κάθε χώρα. Γιατί αυτό δημιουργεί ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ο όγκος αναφορών δεν ανταποκρίνεται αναγκαστικά σε, αυτό το οποίο δίνεται ως δυνατότητα στους πολίτες να ενασκούν το δικαίωμά τους. Με άλλα λόγια, είναι ένα θεμητό πλαίσιο ευνοϊκό πλαίσιο για να μπορέσουμε να εργαστούμε για την ε, ε, αντιμετώπιση αυτών των αναφορών, να ξέρουν οι πολίτες τι σημαίνουν αυτές οι αναφορές και τι μπορεί να γίνει από αυτές, για να μην υπάρξει απογοήτευση σε σχέση με πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν και για να ξεπεράσουμε σε πολλές περιπτώσεις ε, το δυναμικό εργασίας, το, τις δυνατότητες εργασίας που υπάρχουν. Και τούτων λεχθέντων είναι πολύ σημαντικό να το θέσουμε ως θέμα ευθύνης. Ευθύνης ε, για την ε, ανάπτυξη των εργασιών μας έναντι των πολιτών. Να εγγυηθούμε στους πολίτες ότι όχι μόνο είμαστε εδώ για να προασπίσουμε αυτό το δικαίωμά τους και, για, και πρέπει να το υπερασπιστούμε, αλλά είμαστε εδώ για να βρεθούν λύσεις για τα αιτήματά τους και τις αναφορές τους. Αποτελεσματικά και συστηματικά να εξευρεθούν λύσεις. Όλα αυτά τι σημαίνουν ότι το γεγονός το ότι μπορούμε να είμαστε περισσότερο ή λιγότερο ευέλικτοι ή ελαστικοί ή το να δούμε αν θα εξεταστούν κάποιες ως αποδεκτές, αν θα κριθούν κάποιες αποδεκτές ή όχι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος ανάσκησης του δικαιώματος των αναφορών. Πιστεύω σε αυτό το οποίο σχολιάσαμε πιο πριν στη συνάντηση των συντονιστών ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια συνένεσης και τον καθορισμό μιας θέσης ε, και τοποθέτησης κοινή για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Ευχαριστώ. Thank you very much. And I think that was the... Σας ευχαριστώ πολύ και νομίζω ήταν η τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ λοιπόν να δώσω τώρα πάλι το λόγο στην Επιτροπή. Παρακαλώ να είστε σύντομος. Ξέρω ότι είναι πολλές οι ερωτήσεις. Είναι καλό που να απαντήσετε σε όλους, αλλά σύντομα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω υπάρχει κοινό έδαφος για πολλά θέματα και θα ήθελα σε ένα θέμα να επανέλθω που είναι το θέμα των υποθέσεων παράβασης όπου ε, μάλλον εκεί υπάρχει σχέση ανάμεσα στις αναφορές και τον τρόπο με τον οποίο ισχύει και εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και όλοι θα κερδίζαμε νομίζω εάν ήμασταν πιο συγκεκριμένοι στη διάκριση διαφόρων φάσεων. Καταρχήν υπάρχει το θέμα του κατά πόσο το κράτος μέλος στο κεντρικό επίπεδο έχει εφαρμόσει την οδηγία ή την λόγω νομοθεσία στην εσωτερική του ε, νομοθεσία. Αν έχει μεταγράψει δηλαδή την νομοθεσία. Ένα, πρώτο και κύριο. Και εκεί είναι ξεκάθαρο. Είτε το έχει κάνει είτε όχι. Και αν όχι, πάμε στο δικαστήριο, ώστε το δικαστήριο να αποφασίσει ότι όντως υπήρξε παράβαση. Εκεί που περιπλέκονται τα πράγματα είναι οι υποθέσεις όπου αναφέρθηκαν και κάποιοι ευρωβουλευτές, είναι δηλαδή η μεμονωμένη εφαρμογή δηλαδή από εκπροσώπους της διοίκησης, από υπαλλήλου. Και εκεί έχουμε διάφορα εργαλεία. Έχουμε τα απλά, όπως το Solvit για τις μεμονωμένες υποθέσεις, αλλά εκεί όπου συμφωνώ με κάποιες από τις δηλώσεις που κάνατε, όταν υπάρχει εξακολούθηση σχήμα ή πολλές πολλές περιπτώσεις ε, κακής συγκεκριμένης νομοθεσίας, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα ε, για να φτάσουμε δηλαδή σε όλες αυτές τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές που πρέπει να εφαρμόσουν την νομοθεσία. Νομίζω πως θα ήταν καλή ιδέα όλοι μαζί να αυξήσουμε την πίεση, να εκθέσουμε τα κράτη-μέλη ζητώντας τους να έρθουν στην Επιτροπή από την μόνιμη αντιπροσωπεία τους να μας στείλουν κάποιον και από την κυβέρνηση ώστε να δούμε ότι υπάρχουν ε, σημαντικά προβλήματα εφαρμογής και να εξασφαλίσουμε πώς ε, θα φτάσουμε όντως στις τοπικές ε, αρχές. Αυτό είναι το πιο δύσκολο ζήτημα, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε με αυτή την πολλαπλότητα παραγόντων και φορέων. Δεν θα επανέλθω στο θέμα της αποδοχής, γιατί έχει εξαντληθεί το θέμα για την ώρα και είμαι έτοιμος να συνεχίσω φυσικά τη συζήτηση ε, καθώς θα προχωράει ο καιρός. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι βεβαίω ότι όλοι όσοι χρειάζεται να ε, συζητήσουν εις βάθος τα θέματα ε, θα το δεχτείτε, δηλαδή θα δεχτείτε δηλαδή τέτοιου είδους τηλεφωνήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ενημερώσω ότι όσον αφορά τι κρατη ε, κράτη-μέλη τα οποία εμπλέκονται στις εργασίες ε, της Επιτροπής Αναφορών, ας πούμε σήμερα ο Υπουργός ε, Περιβάλλοντος της Ελλάδας θα έρθει στις 3 το απόγευμα, ο κύριος Γιώπας, και αυτό συμβαίνει τακτικά. Συχνά όταν υπάρχει αναφορά που επηρεάζει, που, που, ναι, που αφορά συγκεκριμένη χώρα, συχνά έρχονται οι υπουργοί και θα το αυξήσουμε αυτό στις επόμενες μέρες και μήνες. Και τώρα με τα χαράς να δώσω το λόγο στην νομική υπηρεσία, τον κύριο Αντώνιο Καγιόλα, τον παλιό μου φίλο από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας ε, συστήσω στους συναδέλφους, τους συναδέλφους μάλλον, της Επιτροπής μου που θα εργα... Η κυρία Άννα Ποστησίλου και τον κύριο Ντανιέλ Βεράου, που θα συνεργάζονται με την Επιτροπή σας, θα είναι παρόντες ε, πάντοτε στις Επιτροπές σας και θα σας βοηθούν ε, στις εργασίες σας. Να σας πω δύο λόγια για την νομική υπηρεσία. Θα είμαι σύντομος, ξέρω πως δεν έχετε πολύ χρόνο. Ε, η νομική υπηρεσία είναι μια γενική διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει δύο βασικούς ρόλους. Καταρχήν να αντιπροσωπεύει το Κοινοβούλιο ενώπιον του δικαστηρίου και των εθνικών δικαστηρίων. Δεύτερον, να συμβουλεύει το σώμα σε νομικά ζητήματα και η νομική αυτή βοήθεια μπορεί να είναι τυπική ή και άτυπη. Θα σας το εξηγήσω αυτό. Όσον αφορά την εκπροσώπηση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η νομική υπηρεσία ε, μπορεί να, φέρει, ε, να κάνει ενέργειες, ε, να κάνει προσφυγή στο Γενικό Δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο Δικαστήριο το, το Διοικητικό, όποτε χρειαστεί. Τώρα, όσον αφορά τον συμβουλευτικό μας ρόλο, εμείς ε, μπορούμε να βοηθήσουμε όλα τα πολιτικά σώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Πρόεδρο, το Προεδρείο, τους κοσμήτορες, αλλά και την Γενική Γραμματεία, τη διοίκηση δηλαδή του Ευρωκοινοβουλίου. Σε, αυτήν την αυτό το συμβουλευτικό μας ρόλο, η νομική υπηρεσία, σύμφωνα με την ομολογία του δικαστηρίου, οφείλει να συντάξει ε, ειλικρινείς, αντικειμενικές και εμπεριστατωμένε νομικές νομοδοτήσει. Είναι αρκετά ανεξάρτητη η νομική υπηρεσία έτσι ώστε να σας δώσει τις πιο ε, βέβαιες νομικές νομοδοτήσεις. Μπορούμε να δούμε ότι το πεδίο της τακτικής νομικής διαδικασίας αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Βέβαια, η νομική υπηρεσία συνεργάζεται σε τριμερείς διαλόγους με την Κομισιόν, με το Συμβούλιο σε, ε, και σε διαφόρων ειδών συνεδριάσεις συμμετέχει. Συνήθως, όπως έλεγα, δίνουμε γραπτές νομικές ε, γνωμοδοτήσεις, ε, ε, τυπικές, επί τη βάση της απόφασης του Προεδρείου του 2008 ε, και επίσης μπορούμε να δώσουμε πολλές άτυπες νομικές συμβουλές, θα έλεγα, ε, στη διάρκεια της ε, κοινοβουλευτικής θητείας. Για μας αυτό ε, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τμήμα της εργασίας μας φυσικά. Τώρα, με την άδειά σα θα ήθελα να συνεχίσω στα γαλλικά την παρουσίαση μου αυτή, διότι θα δώσω μια πολύ σύντομη εικόνα της βασικής νομολογίας όσον αφορά τις αναφορές και τα περισσότερα έγγραφα που έχουμε είναι στα γαλλικά. λοιπόν, οι αναφορές αποτέλεσαν αντικείμενο μιας δεκαριάς υποθέσεων που έχουν προσφύγει που ενώπιον των δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Οι αναφερόμενοι έχουν ασχοληθεί με δύο ειδών αποφάσεις. Πρώτον, αυτές που, αποφάσεις που δεν δέχονται τις αναφορές και τις, ε, το κλείσιμο των παρουσιάσεων των αναφορών τους. Εμείς πάντοτε έχουμε περασπίσει τις ε, αποφάσεις που έλαβε η Επιτροπή σας σε όλες τις υποθέσεις εκτός από μία. Στατιστικά δηλαδή το 90% δικαιωθήκαμε ενώπιον ε, του δικαστηρίου. Ακόμα δύο υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον ε, του δικαστηρίου. Πρόκειται για μια ουγγρική υπόθεση όσον αφορά το, τα ε, δικαιώματα ιδιοκτησίας και μια άλλη υπόθεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με το δημόσιο λειτουργήμα. Για την πρώτη, λοιπόν, τις πρώτες λοιπόν αποφάσεις, δηλαδή τις αποφάσεις που δεν δέχονται τις αναφορές θα σας αναφερθώ στην ε, αναφορά Εγκεμπάουερ εναντί του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πρόκειται για μια υπόθεση του 2007 όπου ε, ε, κατηγόρησε την Επιτροπή ο Ενάγων επειδή δεν δέχτηκε την αναφορά του γιατί θεώρησε πως ε, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ένωσης. Το εν λόγω άτομο θεώρησε πως θα πρέπει να γίνει έλεγχος της δικαιοδοσίας και ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής που δηλώνουν ως αποδεκτές τις αναφορές μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγής σε προσακύρωση το δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Αναφορών λόγω ανεπάρκειας ε, και ε, αιτιολόγησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δικαστήριο θεώρησε πως μια τέτοια απόφαση θα πρέπει σαφώς να αναφέρει τα αίτια που δικαιολογούν την κατάταξη αυτής της αναφοράς ως ε, μη αποδεκτής. Πράγμα το οποίο δεν είχε γίνει για την απόφαση αυτή η Αυτή η νομολογία επιβεβαιώθηκε και με άλλα αποφάσει, όπω βάρω έναντι Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλη μια υπόθεση του 2010, J έναντι Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ο ενάγων είναι ανώνυμος. Ε, και εδώ οι προσφυγές απερίφθησαν γιατί σύμφωνα με το δικαστήριο το Κοινοβούλιο σεβάστηκε αυτήν την πλήρη αιτιολόγηση και επιστήνω την προσοχή σας σε αυτό το θέμα της ε, αποδοχής των αναφορών γιατί θα βρείτε πολλές υποθέσεις που έλαβαν υπόψη την ομολογία Πάουερ που επιμένει όπως είπα στην ανάγκη ε, παρκούς αιτιολόγηση. Δεν σημαίνει μακρινά η αιτιολόγηση, αλλά εν πάση περιπτώσει να είναι σαφή, ξεκάθαρη ε, για ποιο λόγο δεν δέχεστε μια αναφορά. Δεύτερη κατηγορία αποφάσεων είναι αυτές που κλείνουν την εξέταση, κλείνουν μια αναφορά. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε την υπόθεση Σονμπέργκερ. Υπάρχουν διάφορες υποθέσει ε, υποθέσεις Σονμπέργκερ εναντίον του Κοινοβουλίου του 2011, η οποία απόφαση θεωρήθηκε αποδεκτή από τη δική σας, ε, η αναφορά μάλλον θεωρήθηκε αποδεκτή από την Επιτροπή σα, ωστόσο... Ε, έκλεισε η αναφορά και διαβιβάστηκε στη Γενική Διεύθυνση που είναι υπεύθυνη για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το δικαστήριο ε, ε, πέριψε ε, αυτή την απόφαση γιατί θεώρησε πως οι αποφάσεις αυτού του είδους δεν μπορούν να προσβληθούν. Η συνέχεια που δίνει ένα κοινοβούλιο, το κοινοβούλιο σε μια αναφορά που θεωρεί αποδεκτή, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των δικαστών της Ένωσης. Το Κοινοβούλιο έχει απόλυτα, απόλυτη διακριτική ευχέρεια πολιτική, έκφρασης πολιτικής άποψης. Είστε απόλυτα ελεύθεροι χωρίς να δώσετε συγκεκριμένη αιτιολόγηση, να το κλείσετε το θέμα. Εδώ είναι δική σας, δικό σας θέμα. Αυτή η ερμηνεία λοιπόν του δικαστηρίου επικυρώθηκε πρόσφατα στην, ε, στην ε, απόφαση που δόθηκε ε, στην υπόθεση Λομνίτσι που ήταν πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ουγγαρίας και του Κοινοβούλιου. Είναι μια υπόθεση του 13. Εδώ ο αναφέρον αμφισβήτησε το δικαίωμα της Επιτροπής να κλείσει την αναφορά βασιζόμενο στην ε, ε, νομολογία ε, Σον Μπέργκερ. Δεν δέχτηκε τον την προσφυγή του κ. Μνίτση. Δηλαδή το Κοινοβούλιο κέρδισε εδώ. Τέλος, να σας πω δύο λόγια για τις σημαντικές αναφορές που αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Μετά από την υπόφαση Σον Μπέργκερ, ο αναφέρον ε, προσεφήγε και πάλι στο δικαστήριο το 2013 τον Ιούλιο. Εκεί ο Γενικός Εισαγγελέας Γιάσκινεν ερμήνευσε τις διατάξεις σε σχέση με τις αναφορές και τη διαδικασία ε, επεξεργασίας των αναφορών να διευκρινίσω ότι το δικαστήριο δεν οφείλει να ακολουθήσει τα συμπεράσματα των γενικών εισαγγελέων αλλά ότι εν γέννη αυτό κάνει στο 90% των υποθέσεων. Ο Γενικός Εισαγγελέας Γιάσκινεν λοιπόν αποφάσισε να ότι μπορεί επισήμως να φέρει γνώση του Κοινοβουλίου ορισμένα θέματα η Επιτροπή Αναφορών χωρίς ο αναφέρον να μπορεί άμεσα να απαιτήσει νομική προστασία. Δεν πρόκειται λοιπόν για ένα ατομικό δικαίωμα το οποίο στόχο έχει ε, νομικές επιπτώσεις ε, σε σχέση με την προσωπική κατάσταση ενός αναφέροντα, αλλά πρόκειται για ένα πολιτικό μέσο, πολιτικό εργαλείο συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή. Το επαναστατικό ε, στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η νομολογία του Power και η, άρα δηλαδή η προσφυγή για ακύρωση δεν, δεν θα μπορεί πλέον να γίνει όποιο, όποιο και είναι το περιεχόμενο αυτής έναντι της Επιτροπής Αναφορών. Αν λοιπόν το δικαστήριο ακολουθήσει την πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα είναι, θα είναι προς όφελό σας γιατί η δική σας γνώμη πάλι θα ισχύει χωρίς τόση αιτιολόγηση και για θέματα αποδοχής ή όχι τη κάθε αναφορά. Θα πρέπει πράγματι να σκεφτόμαστε, να έχουμε υπόψη μα ότι στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων υπάρχει ε, το άρθρο που προβλέπει το δικαίωμα τη αναφορά. Είναι ένα από τα πρωταρχικά δικαιώματα τη Ένωση, δηλαδή το δικαίωμα στην αναφορά. Και σε αυτά θα σταματήσω. Είμαι στη διάθεσή σα ε, για να απαντήσω σε ερωτήσει και αν πάντοτε θα είμαστε στη διάθεσή σας ολόκληρη υπηρεσία μας για να σας βοηθήσουμε στις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ σας ευχαριστώ και επειδή ο χρόνος μας τελειώνει νομίζω θα πρέπει σοβαρά να λάβουμε υπόψη αυτή την προσφορά, να συζητήσουμε περαιτέρω με τις νομικές υπηρεσίες και εγώ προσωπικά εξ ονόματος της Επιτροπής θα συνεργαστώ στενά μαζί σας στις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα νομίζω πως πρέπει να προχωρήσουμε πολύ σύντομα στην αναφορά 0454-2009 της Wendy Clark και θα της δώσω αμέσως Μάλλον, θα δώσω το λόγο στον κύριο Τεμπρόκα που είναι σήμερα παρόν εδώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αυτή η αναφορά αναφέρεται σε μια καταγγελία που έγινε τον Απρίλιο του 2008 στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν. Τότε, αφού εξετάσαμε την καταγγελία, ε, ε, καταλήξαμε ότι ήταν πολύ ισχνή η πιθανότητα τα ζητήματα εδώ να αποτελούν όντως παράβαση ε, των κανόνων ανταγωνισμού της Ένωσης. Συναντήσαμε τον αναφέροντα, ε, εκφράσαμε την εκτίμησή μας και η καταγγελία αυτή αποσύρθηκε τον Ιούνιο, το Μάιο μάλλον του 2008. Δηλαδή λίγες μέρες κράτησε αυτή η αναφορά, έκλεισε τον Ιούνιο του 2008 για μας. Έκτοτε δεν είχαμε καμία επαφή άμεση με τον αναφέροντα, δεν προσπάθησε ξανά να έρθει σε επαφή μαζί μα ή να ζητήσει παραπάνω πληροφορίες ή να καταθέσει κάποια ανεπιπλέον καταγγελία. Για μας είχε κλείσει το θέμα. Ε, όμως, όπως συχνά κάνουμε με τους ε, αναφέροντε, είχαμε υπόψη μας, μάλλον ενημερώσαμε τον αναφέροντα ότι είχε και άλλη νομική οδό μπροστά του, ανοιχτή, αν ήθελε να προσυνεχίσει, ή με την Εθνικές Αρχές ε, ανταγωνισμού γιατί τα θέματα τα οποία ανέφερε ήταν πολύ τοπικής φύσης ε, και η άλλη δυνατότητα ήταν να, έρθει σε να, να, προσφύγει στην ε, δικαιοσύνη του κράτους. Οι τοπικές αρχές κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα με εμά, ότι δηλαδή δεδομένε της φύσης, του, πολύ τοπικής φύσης του θέματος ε, δεν θα βρίσκαμε παράβαση του ανταγωνισμού. Και άρα λοιπόν η Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού ε, έκλεισε την έρευνά του. Της. Δεν, είχα, δεν είχα δεν ήξερα αν ο αναφέροντας όντως είχε προσφύγει δικαστικά για να... στην, στην, στην Εθνική Εισαγγελία. Για μας λοιπόν η έρευνα αυτή, η αναφορά αυτή είχε κλείσει πριν από έξι χρόνια και δεν είχα κανένα νέο έκτοτε. Right uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Τα τελευταία νέα είναι η επιστολή της αναφέρουσας που σας διανέμεται τώρα μόλις έφτασε σήμερα το πρωί και προσωπικά πιστεύω και σε διάλογο με την γραμματεία ότι τα όσα θέλει η αναφέρουσα είναι να ενθαρρύνουμε εμείς τις σκοτσέζικες ε, αρχές να αναλάβουν μια διαδικασία διαμεσολάβησης και μετά να κλείσουμε την αναφορά. Οπότε θα στείλουμε μια επιστολή στη Σκοτία να ενθαρρύνουν την ε, διαδικασία διαμεσολάβησης και να κλείσουμε την αναφορά. Εντάξει, συμφωνείτε, πολύ ωραία. Χωρίς μικρόφωνο. Ωραία, λοιπόν, θα στείλει σχετική επιστολή η γραμματεία στον αναφέροντα. Τώρα, δεν θέλουμε να είναι αναμένο το web stream, γιατί η επόμενη αναφορά είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα. Και ε, ο αναφέρον είναι εδώ στην αίθουσα που βρίσκεστε. Καλώς ορίσατε. Να δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο σε εσάς ε, εξ ονόματος της πλατφόρμα por la defensa de